Dear President, So, die Sitzung ist hiermit wieder. Λοιπόν, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Τα πρακτικά της χτεσινής συνεδρίασης ε, και τα σχετικά κείμενα είναι στη διάθεσή σας. Υπάρχει κάποια αντίρρηση. Όχι. Οπότε εγκρίνονται τα πρακτικά. Πρώτο σημείο στην ενεργησία διάταξη έχουμε